15 λεπτά το πολύ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω σε εσάς, τους ερετούς εκπροσώπους των Ευρωπαίων το ότι ήμουν και εγώ δύο φορές ευρωβουλευτής σημαίνει πως δεν χρειάζεται βεβαίως να μου υπενθυμίσετε την σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν αναλάβω τελικά τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνεργαστώ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ενισχύσω την πολιτική μας πρωτοβουλία και τη δημοκρατική νομιμοποίηση των προτάσεών μας. Η... Τα χαρτοφυλάκια μου είναι το ευρώ και ο κοινωνικός διάλογος. Θεωρώ λοιπόν πως τα καθήκοντά μου είναι η προώθηση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σταθερότητα, συντονισμός της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και βεβαίως στενότερη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, γεννήθηκα και μεγάλωσα πίσω από το παραπέτασμα. Για 50 χρόνια η Λετωνία δεν μπορούσε να είναι μέρος της Ευρώπης, δεν είχαμε βασικά δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες. Πριν από 25 χρόνια έπεσε το μου παραπέτασμα και έτσι άνοιξε ο δρόμος για ειρηνική δημοκρατική αλλαγή στην Ήπειρό μας. Η προοπτική για χώρες όπως η Λετωνία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή η οποία αποτελεί στο θεμέλιο της δημοκρατικής, οικονομικής και κοινωνικής μεταμόρφωσης. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω στην δύναμη του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Πιστεύω στις βασικές ευρωπαϊκές αξίες της δημοκρατίας, της κοινωνικής οικονομίας αγοράς και των ίσων ευκαιριών. Μόνο μαζί θα, μπορούμε, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ενός κόσμου που αλλάζει γρήγορα, της παγκοσμιοποίησης, της γύρανσης και της κλιματικής αλλαγής. Είχα την τιμή να είμαι πρωθυπουργός Λετωνίας σε τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις από το Μάρτιο 2009 μέχρι και φέτος τον Ιανουάριο. Έλαβα καθήκοντα όταν η χώρα μου περνούσε την βαθύτερη οικονομική κρίση εντός της Ένωσης. Προτεραιότητα να αποκατασταθεί η ανάπτυξη και οι θέσει εργασία ε, το συντομότερο δυνατόν. Ως αποτέλεσμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, η Λετωνία βγήκε από την κρίση και έγινε μία από τις οικονομίες της Ευρώπης που αναπτύσσεται ταχύτερα. Υπήρχαν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, κυρίως ε, τα οικονομικά κίνητρα μέσω της ε, επιτάχυνσης της χρήσης των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων και δημιουργήσαμε ένα επιπλέον δίκτυ ε, κοινωνική ασφάλισης. Επίσης εκπληρώσαμε τα κριτήρια του Μάστριχτ και ενταχθήκαμε φέτος στο ευρώ. Αυτές οι διαδικασίες δεν θα ήταν δυνατόν να λάβουν χώρα χωρίς έναν διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους για τις ευαίσθητες πολιτικές και κοινωνικές αποφάσεις προετοιμαζόμενοι για την υιοθέτηση του ευρώ τη στιγμή που υπήρχε κρίση στην ευρωζώνη επιδείξαμε την εμπιστοσύνη μας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και το ευρώ τη στιγμή που άλλοι το αμφισβητούσαν. Στο παρελθόν ήμουν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος του ε, Λετωνικού Κοινοβουλίου, Υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής οικονομολόγος της Κεντρικής Τράπεζας. Θεωρώ πως η εμπειρία μου αυτή μου δίνει την απαραίτητη γνώση για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι μπορώ να συνεισφέρω σε στην κοινωνική, οικονομική και νομισματική πολιτική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΟΝΕ και να διατηρήσουμε τη σταθερότητα του ευρώ, να εργαστούμε προς μια σύγκληση οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών με τις πολιτικές της αγοράς εργασίας. Εάν με εγκρίνεται λοιπόν στη θέση αυτή, θα εργαστώ σκληρά για να διαβασφαλίσω πως οι στόχοι της σταθερότητας του ενιαίου νομίσματος και της μακροοικονομικής διακυβέρνησης θα συμβαστούν με την κοινωνική δικαιοσύνη και την συμπερίληψη όλων. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να αντιμετωπίσει τη χειρότερη κρίση στην ιστορία τη και να διαφυλάξει το ενιαίο τη νόμισμα. Αυτή τη στιγμή όμως ε, προβλέπεται πως τα επόμενα 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτυχθεί με ένα 1,5% τα επόμενα 10 χρόνια όπως είπα. 1% λιγότερο δηλαδή από ό,τι στην προηγούμενη δεκαετία. Η κρίση εξακολουθεί λοιπόν να πλήττει τις κοινωνίες μας. Ε, στην Ευρωζώνη είναι πάνω από 11% η ανεργία, στους νέους είναι πάνω από 20% και 16% των Ευρωπαίων μεταξύ 15 και 29 δεν είναι ε, δεν έχουν ούτε δουλειά ούτε εκπαιδεύονται. Η Ευρώπη δεν μπορεί να χάσει μια ολόκληρη γενιά. Όλοι ξέρουμε πως ε, η κρίση αυτή δεν ήταν μια απλή μείωση των οικονομικών μεγεθών. Ε, οι αιτίες της ήταν αδυναμίες στις οικονομικές μας δομές. Γι' αυτό πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο με έναν πληθυσμό που γυράσκει με υψηλό επίπεδο χρέους και πολύ, χαμηλή, ε, πολύ χαμηλό πληθωρισμό η Ευρώπη να περάσει σε μια περίοδο χαμηλής ανάπτυξης ή ακόμα και στασιμότητας. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους και να επανέλθουμε στο κατεύθυνση της αηφόρου ανάπτυξης. Οπότε χρειάζονται να αναλυθούν συγκεκριμένα και συντονισμένα μέτρα και από την πλευρά τη ζήτηση και τη προσφορά και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει οι προτάσει τη Κομισιόν να μεταφραστούν γρήγορα σε έργα. Αφετηρία θα είναι το επενδυτικό πακέτο 300 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων τα επόμενα τρία χρόνια και εδώ πέρα βέβαια συγκεκριτικό ρόλο θα παίξει ο αντιπρόεδρο για δουλειέ και ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Χρειάζεται λοιπόν επενδύσεις υψηλή ποιότητα για να διατηρήσουμε την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και για την υφιστάμενη χρηματοδότηση. Τα ευρωπαϊκά Διελευθερωτικά ταμεία πρέπει να επενδύονται σωστά και πρωτοβουλίε όπω η εγγύηση για την νεολαία πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Η κρίση κατέδειξε ότι υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες στον αρχικό προγραμματισμό του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου. Τα τελευταία χρόνια ελήφθησαν σοβαρά βήματα για την αντιμετώπιση τους. Η ε, δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρνηση ενισχύθηκε. Επίσης ορίστηκε ένα πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης και υπάρχει μια εξάντε, ένας συντονισμός των εθνικών πολιτικών που ενισχύθηκαν υπό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Επίσης, ορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα ανάσχεσης τα τελευταία χρόνια. Η Τραπεζική Ένωση έχει καταλήξει και οι αδυναμίες των ισολογισμών των τραπεζών θα πρέπει να μας οδηγήσει σε συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να συνεχίσει η δανειοδότηση στην πραγματική οικονομία. Σήμερα είμαστε, η ευρωπαϊκή οικονομία είναι πολύ πιο εύρωστη και μπορεί να οδηγήσει σε ένα πραγματικά ανταγωνιστικό πλαίσιο και ένα πλαίσιο που δεν προβαίνει σε κοινωνικούς αποκλεισμούς. Επίσης θα πρέπει να έχουμε έναν ευρύ κύκλο πολιτική συντονισμού το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έτσι ώστε να ορίσουμε συνεκτικές πολιτικές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το βαθμολόγιο απασχόλησης και κοινωνικών δικτών. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόσουμε την ευελιξία που ήδη υπάρχει του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας. Θα πρέπει να έχουμε ίση μεταχείριση, να διασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών και διαχείριση κατά διαφανή τρόπο. Ο οικονομικός διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί. Έχουν γίνει σοβαρά βήματα μέσα στα πλαίσια της ενίσχυσης ε, του χώρου του ευρώ μέσω του, του pac και του 6 pac Εάν διοριστώ από το σώμα σας, θα αναλάβω όλα τα μέτρα έτσι ώστε να ενισχύσω αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την σταθερότητα και την αξιοπιστία μας μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών επιπτώσεων των πολιτικών μας. Παράλληλα θα πρέπει να βελτιώσουμε την εφαρμογή των συγκεκριμένων συστάσεων προς τα κράτη-μέλη θεωρώ ότι θα πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα έτσι ώστε να έχουμε υψηλότερο επίπεδο η οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. Θα πρέπει να μειώσουμε την ε, αδιαφάνεια στον τομέα των εισοδημάτων και την ανισότητα καθώς και τη φτώχεια. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την ε, ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Αγαπητά μέλη, πιστεύω ότι η μελλοντική ανάπτυξη της ΟΝΕ αποτελεί έναν άμεσο αλλά και μεσοπρόθεσμο στόχο όπως ορίστηκε από το προσχέδιο για μια πραγματική και αυθεντική ΟΝΕ. Έτσι θα μπορέσουμε να ε, προωθήσουμε την ΟΝΕ με βάση αυτά τα δεδομένα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε στο μέτρο του δυνατού και να συμπεριλάβουμε στη συνεργασία αυτή και τα 28 κράτη-μέλη ο χώρος της Ευρωζώνης θα πρέπει να μείνει ανοιχτό σε νέα μέλη εάν πληρούνται τα κριτήρια του Μάστριχτ. Υπό αυτή την έννοια χαίρομαι διότι η Λιθουανία θα γίνει το 19ο μέλος της Ευρωζώνης στους επόμενους τρεις μήνες. Αυτό αφορά βέβαια και τη χρήση της κοινοτικής μεθόδου. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις διάφορες επιλογές λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και την ενδεχόμενη αλλαγή των συνθήκων. Αγαπητά μέλη, και αν διοριστώ αντιπρόεδρος, η εντολή μου θα αφορά μία εργασία για την επανεξισορρόπηση των ε, όρων σταθερότητας μέσα στα πλαίσια των χωρών της ε, Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ε, δέχομαι τη δέσμευση του Προέδρου Γιούνκερ μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής συνεργασίας και αποτίμησης. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί κράτη-μέλη να προστρέξουν σε τέτοια προγράμματα πλέον. Τη στιγμή που ορίστηκε η Τρόικα και διορίστηκε για να διαχειριστεί μια κατάσταση οικονομικής καταστροφής θα πρέπει στη συνέχεια να, να, να αντικατασταθεί από νέα νόμιμα δημοκρατικά μέσα και διαρθρώσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και να ασχοληθούμε και με τις δύο πλευρές του νομίσματος, δηλαδή το οικονομικό σκέλος και το κοινωνικό. Διαμέσω της ιστορίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και κοινωνικού διαλόγου ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε ε, ανταλλαγές απόψεων με τους κοινωνικούς εταίρους επί της ουσίας. Ο κοινωνικός διάλογος είναι απόλυτα αναγκαίος έτσι ώστε οι μεταρρυθμίσεις να καταστούν δυνατές και βιώσιμες. Είναι ένα απαράβατος όρος για την ευημερία της ΟΝΕ. Θα συνεργαστώ με τους Επιτρόπους Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και κινητικότητας ε, της αγοράς για να ενισχύσουμε αυτά τα μέτρα και σε εθνικό επίπεδο. Ο ρόλος ε, του Αντιπροέδρου για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο αποτελεί απάβγασμα του στόχου του Προέδρου για την ενίσχυση του ρόλου του κοινωνικού διαλόγου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την άμεση συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίζομαι στην υποστήριξή σας για να προωθήσω την οικονομική και, κοινωνικό, και κοινωνική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.